Παρακαλώ κύριε Ντομένιτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χθε στη Φλωρεντία συνέβη ένα πολύ σοβαρό γεγονός το οποίο προκαλεί φρίκη και αγανάκτηση. Ένας πενιντάρης ένοπλος πυροβόλησε σε δύο αγορές στην, μάλλον δύο και σκότωσε δύο Σενεγαλέζους ε, πολιτές ο δολοφόνος ε, μετά αυτοκτόνησε πρόκειται για έναν άκρο δεξιό ρατσιστή που θα ήθελε να δολοφονήσει άτομα άγνωστα και τα οποία ήταν ε, στα θύματα μάλλον του χρώματος του δέρματός Στο παρελθόν υπήρξα για 10 ε, χρόνια δήμαρχος της ε, Φλωρεντίας. Είναι μια πόλη ε, αντιστασιακή. Στην Φλωρεντία λοιπόν στέβει αυτό το ρατσιστικό έγκλημα το οποίο καταδεικνύει ότι η ναζική και η φασιστική τρέλα μπορεί να εκδηλωθεί απανταχού και δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι την έχουμε ε, εξαλείψει. Κύριε Πρόεδρε, σα ζητώ να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επαναλάβουμε τη δέσμευση αυτού του σώματο κατά κάθε μορφή ρατσισμού και ε, ξενοφοβία και του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων των, α, απανταχού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ντομένιτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και υπενθυμίζω πως σήμερα το πρωί ε, με την έναρξη της συνεδριάσεώς μας ο πρόεδρος Μπούζεκ ήδη έκανε δηλώσεις ε, πολύ αυστηρές σε σχέση με τα όσο συνέβησαν τόσο στη Φλωρεντία όσο και αυτά που συνέβησαν στην Λιέγη. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε τα συναισθήματα και τα λόγια καταδίκης που εξέφρασε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια ο κύριος ε, Μπούζεκ. Τώρα και τώρα περάσουμε Έκθεση Αλμπερτίνη σχετικά με το μηχανισμό πρωταξιακής βοήθεια. Άρχεται ψηφοφορία. Avete tutti? Ψήφισαν άπαντες. Βιαστείτε παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία. Ενεκρίθημε με στην τριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Αλμπερτίνη, έκθεση Περέγιο Ροντρίγκε. Ονομαστική ψηφοφορία στο πρώτο μπλοκ του τροπολογίου. Άρχιε ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρα τη ψηφοφορία. Ενεκρίθησαν. Τώρα ψηφίζουμε με ορμαστική ψηφοφορία στην τροποποιημένη πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Συντηρητική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρα της ψηφοφορίας. Και εδώ συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Σεγίτα έκθεση Νιούτον Ντάν. Το πρώτο μπλοκ των ψηφί πέρουν. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η πρόταση της Επιτροπής ε, με την τροποποίηση που εδέχθηκε ψηφί πέρα κατά αποχές ε, δεκτή. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, την ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, πέρα ψηφοφορίας. Συντριπτική και εδώ η πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Έκθεση Χάγκλουμ για τη Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι κάπως ασυνήθιστη αυτή η διαδικασία ψηφοφορίας για την έκθεση αυτή, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η διαδικασία ψηφοφορίας θα έχει ως εξής ψήφος υπέρ της έκθεσης σημαίνει ότι συνενούμε στην παράταση του πρωτοκόλου. Ενώ αν ψηφίσουμε κατά σημαίνει ότι δεν συνενούμε προ την παράταση του πρωτοκόλου διότι δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε τροπολογίε. Σύμφωνα με την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ανάπτυξη, αυτό ήταν ψήφο κατά, ενώ η Επιτροπή Αλληλεία, παρά τη δική μου εισήγηση, αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ. Αυτό ήθελα να πω προ διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τι διευκρινήσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Bene. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πρόταση απόφαση σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Έκθεση Μπόλσου. μυστική ψηφοφορία. Είσαστε παίοντες, δεν έχετε ανάγκη από οδηγίες, θα έχετε το μπλε φωτάκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Έληξε ψηφοφορία. Με συντριπτική πλειοψηφία εξελέγεται το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τώρα περνάμε στα τέσσερα ψηφίσματα για την Συμφωνία Ελευθερική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βασιλείου του Μαρόκου. Πρόταση ψηφίσματο ε, η πρώτη είναι άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έληξε ψηφοφορία. απορρίπτονται οι τροπολογίες και το ψήφισμα απορρίπτεται τώρα το ψήφισμα των πρασίνων ε, και των φιλελευθέρων δεν τροπολογία ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται πρόταση ψηφίσματος ε, τριών πολιτικών ομάδων ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκρατών Γιάλτε ε, ψηφίπερ. Α, συγγνώμη, υπάρχει μια τροπολογία. μόνο τέσσερα Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 4. Μετά την παράγραφο 7, ε, ο κύριος ε, Γκουίντο Μιλάνα προτείνει μια φορική τροπολογία. Κύριε Μιλάνα, μπορείτε παρακαλώ να μας εκθέσετε την τροπολογία σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία η ε, οποία θέλει να θέσει στο κείμενο αυτό τον όρο των ε, Σεβασμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κείμενο έχει εξή. Μετά από το σημείο 7 του ψηφίσματο. Ε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει στην συμφωνία με το Μαρόκο την ρήτρα του Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κοινωνικούς κανόνες και σε όλες τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Νομίζω ότι αυτή η τροπολογία βελτιώνει το ψήφισμα και δίνει μια σαφή ένδειξη προς την Επιτροπή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων να λάβει λοιπόν υπόψη της ότι στον χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, συχνά το, για τα θέματα αυτά το Κοινοβούλιο είναι διχασμένο. Λοιπόν, υπάρχουν ενστάσεις από πλευρά συναδέλφων, ε, δεν υπάρχουν ενστάσεις και διαφωνίες, ζητώ να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Ο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, ο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη και σε κάθε εμπορική συμφωνία που συνάπτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι δεν είναι. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακριβές αυτό το οποίο προτείνει ο κ. Μιλάνα. Ma eh, io penso Νομίζω ότι δεν ε, αποτελεί επικάλυψη ούτε επανάληψη πρώτος κ. Μιλάνου. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό είναι να προσθέτουμε και να μην αφαιρούμε. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία του κύριου Μιλάνα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρα ψηφοφορίας. Συντριπτική πλειοψηφία. Η τροπολογία έγινε δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες. Έληξε η ψηφοφορία. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πρόλεση ψηφίσματος, ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Και εδώ μεγάλη πλειοψηφία υπέρ. Σε χαρακτήρια κύριε Σιγητά. Περνάμε στην έκθεση Λίζεκ. Ο εισηγητής ε, ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πιο δυσηγητές για τη συνεργασία τους και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν ε, στην ε, κατάρτιση του εγγράφου το οποίο ψηφίζουμε μέσα σε μια δύσκολη δημοσιονομική κρίση. Αλλά υπενθυμίζουμε μια βασική αρχή όπως αυτό της ασφάλειας και γι' αυτό προτείνω να υπερσυζητηθεί η έκθεση. Ψηφίζουμε τροπολογίες 1 και 2 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Δεκτές. Παράγραφος 3 χωριστά. μένουμε νομιστική ψηφοφορία και τα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, την ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα είναι δεκτό. Δεύτερο τμήμα, την ψηφοφορία. Ψήφισαν απαντές. της ψηφοφορίας. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 5. Ε, πρώτο τμήμα. άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν απάντες. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. Παράγραφος 10. Πρώτο τμήμα. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. 23. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 29. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Παράγραφος 35. Άρχη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 36 υπέρ. Συγγνώμη, άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτεί. 37. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτεί. 38. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 40 υπέρ. Συγγνώμη, άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν σε έληξη ψηφοφορία. Δεκτή 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Δεκτή. 59. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 60 χωριστά το πρώτο τμήμα άρχιτε η ψηφοφορία έληξε το πρώτο τμήμα έγινε δεκτό απορρίτερη συγγνώμη απερίφθη το δεύτερο τμήμα άρχιτε η ψηφοφορία σε έληξε ψηφοφορία δεκτό το δεύτερο τμήμα 70 ψηφίζουμε Έληξη ψηφοφορία. Δεκτό. 71. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξη. Δεκτή. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Συντηρητική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Και τώρα περνάμε στην διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Κοινέ προτάσεις ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 15. Το πρώτο τμήμα Διανατάσσεως της χειρός, υπέρ κατά αποχές, ε, δεκτό, δεύτερο τμήμα, την ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρα ψηφοφορίας. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 16, χωριστά. Ονομαστική. Όχι, για το πρώτο τμήμα με διανατάσσεως της χειρός, ψηφί Κατά, αποχές ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτό το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 1. Χωριστά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε. Συγγνώμη γιατί δεν είδα τα χέρια. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο του κοινού ψηφίσματος ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτό Πρέπει να διακόψουν τις ψηφοφορίες διότι έχουμε την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Θα συνεχίσουμε μετά το πέρας της τελετής.